προφανώς σε κάποιες περιπτώσεις αποκαλύπτουν βαθιά συναισθήματα. Προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Αυτό αναγνωρίζεται, πιστεύω, από τον τελευταίο μιλήτη, και τον κύριο Λόπες Αγγιγιάρ και τον κύριο Ντεπρέ προηγουμένω. Προσπαθήσαμε να καλύψουμε κάποια θέματα που έθιξαν οι ομάδες απόψε. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα ενισχυμένο από τον έλεγχο και την τροφοδοσία των απόψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Την χάνει υποστηρίξεω στο Συμβούλιο, άρα δεν είναι κατά των κρατών μελών. Αλλά πιο σημαντικό για μένα έχει τη στεναρή υποστήριξη εκείνων που στην πρώτη γραμμή. Ε, έχει την υποστήριξη των αστυνομικών, των συνοριοφυλάκων, των αξιωματούχων, των υπεύθυνων για τη μετανάστευση, που πρέπει να κάνουν τη δουλειά του, δηλαδή να μα ε, προστατεύουν και να μα κρατούν ασφαλεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα οι δύο εισηγητέ. Πρώτα απ' όλα Λένας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι αλήθεια ότι από την αρχή αυτή της διαδικασίας πέρασαμε πάρα πολλές ώρες να συζητάμε στο Κοινοβούλιο με την Επιτροπή για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε, τι μπορούμε να βελτιώσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Και όλη αυτή η δουλειά νομίζω καρποφόρησε. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους εδώ, οι οποίοι εξέφρασαν τη στήριξή τους στην πρόταση. Νομίζω ότι περισσότεροι από εμά στηρίζουν την πρόταση. περισσότεροι από εμά είπαν ότι υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ε, τα ακούσαμε και πριν, ναι, ναι δεν πρόκειται για δύο στοιχεία τα οποία είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Όχι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις και είναι καλά νέα αν κάποιος νοιάζεται για την καταπολέμηση της απάτης όσον αφορά της ταυτότητας, αν νοιάζεται κανείς για την πολιτική μας ασφάλεια προκειμένου αυτή να είναι πιο αποτελεσματική και είναι θετικό αν θέλουμε η αστυνομική μας, η ε, τελωνιακοί μας, οι συνοριοφύλακοί μας να έχουν τα κατάλληλα εργαλεία για να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και βοηθάει πολύ νομίζω και εν ώψη των ευρωεκλογών όπως το είπε και κάποιος νωρίτερα. Αν βέβαια δεν μας ενδιαφέρει η ασφάλεια, η καταπολέμηση της απάτης κτλ, εντάξει, μπορεί κανείς να ψηφίσει για τους πρασίνους ή για την ε, άκρα αριστερά. Ευχαριστώ. Και τώρα ο Σάρφος Μέλου. Λοιπόν, κλείνοντας να πω ότι αναφερόμενοι στις αρχές, στις αστυνομικέ δυνάμεις που καθημερινά δικαινεύουν τη ζωή τους για να εγγυηθούν την ελευθερία μας, για αυτές τις αστυνομικέ δυνάμεις και για τους άλλους φορείς, τους αρμοδίους, πρέπει να βρούμε τις καλύτερες απαντήσεις, Europol, Frontex, EISA, η υπηρεσία αλλοδαπών και διάφορες άλλες αρμόδιες υπηρεσίες της χώρας μου. Δεύτερο σχόλιο, αντίθετα με αυτά που είπαν οι πράσινοι και οι κομμουνιστές, οι πράσινοι μας λέγουν ότι με αυτό το σύστημα εμείς ελέγχουμε τους εγκληματίες αλλά και τους ε, αθώους πολίτες. Αυτό είναι σύνηθες. Αν ξέραμε ποιοι θα ήταν οι εγκληματίες δεν θα κάναμε έρευνες. Διότι Όλος ο κόσμος είναι ανάμεικτος, λοιπόν, ε, πρέπει να ερευνήσουμε εκεί, πρέπει να διεξάγονται έρευνες, ούτως ώστε οι, οι αθώοι που οι περισσότεροι ευτυχώς είναι αυτοί, ε, ε, διαχωρίζονται από τους εγκληματίες και έτσι μπορούμε να καταπολεμούμε την τρομοκρατία και να εγγυηθούμε επίσης την εύρυθμη λειτουργία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να απαντήσω σε, στους κομμουνιστές που ανησυχούν για τα θέματα της νομιμότητας θα ήθελα να τους πω ακόμα και αν έχουν αποχωρήσει διότι η συζήτηση φαίνεται δεν είναι αρκετά σημαντική για αυτούς. Θέλω να πω λοιπόν εμείς ότι θέλουμε να εγγυηθούμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα κινηθούμε με το μεγαλύτερο σεβασμό όσον αφορά τα στοιχεία. Θα τα κάνουμε πολύ καλύτερα όλα αυτά από τα καθεστώτα που καταραίουν, από καθεστώτα που βρίσκονται στη Βενεζουέλα, στην Κούβα ή στη Βόρεια Κορέα, όπου δεν γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και συλλέγουν όλες τις πληροφορίες, γίνονται συλλήψεις αυθαίρετες ε, για διαφορά απόψεων, παραδείγματος χάρη που εκφράζεται, ή εξαφανίζεται ε, κόσμος ξαφνικά. Ε, λοιπόν, θέλουμε εμείς να ε, κινηθούμε βάσει τις νομιμότητες και να εγγυηθούμε όμως και την ασφάλεια στον αφορά τους πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε Μέλλου. Ολοκληρώνεται έτσι η συζήτηση. Επόμενο θέμα στη μέση διάταξη. Κοινή συζήτηση. Α, όχι, όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, η ψηφοφορία θα γίνει στη δεύτερη ολόμερα του Απριλίου. Τώρα, το επόμενο θέμα είναι η συζήτηση για την έκθεση της συναδέλφου Νίμπλερ αύξηση αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφαιρεγιότητας και απαλλαγής. Η συγγήτρια. Τέσσερα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ τους Σκιώδης για τη στήριξή τους κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού. Νομίζω ότι η οδηγία για τις προληπτικές αναδιαρθρώσεις δεύτερη και δεύτερη δυνατότητα για τις ε, επιχειρήσεις είναι πραγματικά ένα ορόσημο για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις μας. Ξέρετε Κάθε χρόνο ε, πτωχεύουν 200.000 ε, εταιρείε και χάνονται 1,7 εκατομμύρια θέσει εργασία. 5% των επιχειρήσεων που δημιουργούνται στην Ευρώπη ε, πτωχεύουν μέσα σε 5 χρόνια. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε την επιχειρηματικότητα και αν διευκολύνουμε την αναδιάρθρωση των εταιριών που αντιμετωπίζουν τις χέρειες χρηματοδότηση, τότε κάνουμε κάτι θετικό. Και αν στηρίξουμε τις ε, επιχειρήσεις που δημιουργούνται για πρώτη φορά και που δεν ολοκληρώθηκε καλά την πρώτη φορά η λειτουργία τους και θέλουμε να τις βοηθήσουμε να, τους, ε, να σταθούν και πάλι στα πόδια τους πρέπει να τους δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία γιατί οι νέοι θέλουν χρόνο για να μάθουν πώς να λειτουργούν μια επιχείρηση. Ήταν δύσκολη η αρχή αυτής της ε, διαδικασία. Έχουμε 28 διαφορετικέ θέσει διαδικασίας αναδιάρθρωσης. Σε κάποιε χώρε όπω η Βουλγαρία και η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Κροατία δεν υπάρχουν καθόλου προβλέψει για αναδιάρθρωση. Και σε άλλε χώρε είναι πολύ αυστηρέ προποθέσει όπω η δική μου για παράδειγμα, η Γερμανία. Και υπάρχουν χώρε επίση που είναι χαλαροί όπω η Γαλλία, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλε για την αναδιάρθρωση. Επιπλέον, οι αναδιαρθρώσει ε, βασίζονται σε διαφορετικές νοοτροπίες. Σε πολλές χώρες όπως στη Γερμανία η αναδιάρθρωση για, σε περίπτωση ε, πτώχευσης γίνεται κυρίως με βάση την επιστροφή των χρημάτων στους πιστωτές ενώ σε άλλες χώρες κυρίως ε, προσπαθούν να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας. Με την οδηγία αυτή τι προβλέπουμε για αυτές τις προληπτικές αναδιαρθρώσεις προβλέπουμε μια καλή ισορροπία μεταξύ των διαφόρων αυτών ε, τρόπων λειτουργίας. Έχουμε τρία τμήματα. Πρώτα απ' όλα έχουμε ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που θα πρέπει να δημιουργήσουν τα κράτη-μέλη. Το δεύτερο μεγάλο τμήμα της έκθεσης έχει να κάνει με τις προληπτικές αναδιαρθρώσεις και το τρίτο τμήμα της οδηγίας αφορά την απαλλαγή. Τα ε, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης είναι καλά Πρέπει να υπάρχουν σε όλε τι χώρε, ούτω ώστε να τα χρησιμοποιούν οι επιχειρήσει για να μπορούν εύκολα και εγκαίρω να αποφασίζουν αν χρειάζεται τέτοια αναδιάθρωση. Σε κάποιε χώρε υπάρχουν, σε άλλε όχι. Για την προληπτική αναδιάθρωση τώρα θέλαμε καλύτερη ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων όλων των εμπλεκομένων, πρώτα απ' όλα των πιστωτών και αυτών ε, ε, που χρωστάνε χρήματα. Είχαμε μια καλή πρόταση αλλά κυρίως ε, είχε να κάνει με, το, με τα συμφέροντα των ε, δανειστών, των δανειζομένων μάλιστα, μα ε, καλύτερα θέλουμε με την έκθεσή μας να καταστεί σαφέστερο πώς και τι ρόλο θα παίζουν οι συμμετέχοντες σε αυτή τη διαδικασία προληπτικής αναδιάρθρωσης. Είπαμε, για παράδειγμα, αν υπάρχει κάποιος διαχειριστής και αν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική ή εθελοντική η συμμετοχή ενός διαχειριστή. Αυτό ενδιέφερε πολύ πολλούς συναδέλφους. Και επίσης τους ενδιέφερε ε, η διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους. Ε, καταφέραμε να υπάρξει μια ισορροπία, χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα, πιστεύω ότι εργαστήκαμε πολύ καλά και για την, ε, ε, τον καθορισμό των λεπτομεριών και για την απαλλαγή τα πήγαμε καλά. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει δυνατότητα αυτή η απαλλαγή να γίνει μέσα σε τρία χρόνια. Συνολικά λοιπόν είναι καλό το αποτέλεσμα. Ελπίζω να μπορέσουμε να πείσουμε τους περισσότερους και να βοηθήσουμε και τους επιχειρηματίες να φτιάχνουν επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε Νίμπλερ. Και τώρα ο Επίτροπος Κίνγκ. Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, αυτή η οδηγία που θα ψηφίσετε αύριο έχει δύο στόχους. Θέλει να βοηθήσει τη διάσωση επιχειρήσεων που βρίσκονται υπό οικονομική πίεση και να επιτρέψει επιτρέψει στους τίμιους επιχειρηματίες που απέτυχαν να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτά τα μέτρα θα διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία του κεφαλαίου, όπως επίσης και την ελεύθερη εγκατάσταση επιχειρήσεων. Αλλά θα προσφέρει και μια ευρωπαϊκή προσέγγιση με άρση των εμποδίων που οφείλονται στις διαφορές που ακούσαμε εξαιτία διαδικασιών εθνικής νομοθεσίας όσον αφορά την ε, ε, πτώχευση και την δεύτερη ευκαιρία. Αυτή η νοοτροπία λοιπόν διάσωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντική για να ενθαρρύνουμε την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη. Οπότε, εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια την κυρία Νίμπλερ αλλά και του κοιόδε εισηγητέ για την εξαίρετη συνεργασία και τη σκληρή δουλειά που έκαναν. Η οδηγία αυτή λοιπόν φροντίζει να υπάρχουν προδιαγραφές ενιαίες για την ε, διάσωση ώστε οι επιχειρήσεις που είναι σε δυσκολία να μπορέσουν να περάσουν σε αναδιάρθρωση με συγκεκριμένα πλαίσια και να συνεχίσουν έτσι να λειτουργούν. Επίσης διασφαλίζει ότι οι τίμοι επιχειρηματίες έχουν δεύτερη ευκαιρία ακόμα και αν έχουν πτωχεύσει με απαλλαγή και να μπορέσουν να ε, προβούν σε νέα επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα στα τρία χρόνια. Έτσι λοιπόν αυτές οι διαδικασίες βοηθούν να κερδίσουμε και χρόνο. Θα υπάρξουν επίσης περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης στην εσωτερική αγορά από τις επιχειρήσεις, θα χάνουν ε, θα κάνονται λιγότερες θέσεις απασχόληση, ε, θα βοηθήσουμε να υπάρχουν λιγότερα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και να υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για τους επιχειρηματίες εκείνους που θέλουμε να στηρίξουμε αν χρειάζονται μια νέα αρχή. Ελπίζω αύριο με την ψηφοφορία σας να στηρίξετε την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλβέτ Δύο Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε Βρετανέ, Επίτροπε, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ να ασχοληθείτε με αυτήν την σημαντική πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι ουσιαστικά σημειώνει μια αλλαγή στην οτροπία και στην μεταχείριση που επιφυλάσσουμε στην επιχειρηματική δραστηριότητα και στην ανάληψη κινδύνου στην Ευρώπη. με διαφορά από ό,τι ισχύει στην Αμερική. Κάθε χρόνο πάρα πολλές επιχειρήσεις φτωχεύουν με αποτέλεσμα να χάνονται 7 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Και γιατί, γιατί υπάρχει μια ακαμψία στην εφαρμογή των κανόνων και μια έτσι διοικητικού χαρακτήρα και ε, λογιστικού χαρακτήρα αντιμετώπιση στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως αυτή η νομοθετική πρόταση να προχωρήσει γιατί επηρεάζει απευθείας το πιο σημαντικό στοιχείο της κοινωνίας μας, το ενεργητικό μας, τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους οι οποίοι απασχολούνται από τις επιχειρήσεις αυτές. Τέσσερα πράγματα έχω να πω. Μεγαλύτερη ε, συνοχή Ενία αγορά με περισσότερη αλληλεγγύη και περισσότερη αξιοπιστία και στον οικονομικό κόσμο. Επίσης, διευκολύνει την νομική βεβαιότητα διασυνοριακά, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό για να καταργήσουμε τα σύνορα. Αυτό είναι το μέλλον της Ευρώπης. Επίσης, φροντίζει για την αναδιάρθρωση των βιώσιμων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες Υπάρχει αυτή η προτεραιότητα ε, που έχουμε συχνά να τηρούμε τον νόμο. Ναι, αλλά συγχρόνως πρέπει να προστατεύουμε τους επιχειρηματίες, να δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία και στους επιχειρηματίες και στους εργαζόμενους. να στοιχηματίζουμε περισσότερο στην επιβίωσή τους παρά στην τιμωρία τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω τόσο αλφομάτα, οπότε τρία λεπτά ο κύριος Βόμποντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, συγχαρητήρια στη συνάδελφο Αγγέλικα Νίμπλερ. Είναι έξοχη η έκθεση της. Η προληπτική αναδιάρθρωση είναι βέβαια σημαντικότατη σαν εργαλείο για τους Ευρωπαίους επιχειρηματίες εάν σε όλη την Ευρώπη εφαρμόζουμε τους κανόνες αυτούς, αυτό θα είναι κάτι πολύ καλό για τις ελευθερίες μας. Την ελεύθερια της διακίνησης, την ελευθερία των επιχειρήσεων να κινούνται και να δραστηριοποιούνται και θα στηριχθούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι το 99% των επιχειρήσεων. Και καμιά φορά ή πολύ συχνά δεν είναι πολύ ισχυρέ οικονομικά. Αυτό λοιπόν αποτελεί προστιθέμενη αξία. Ελάχιστη εναρμόνιση. Επίσης, παρέχει επαρκή χώρο, ούτω ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να κινηθούν με κανόνες και να μπορούν να τους εφαρμόζουν ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της πολιτισμικές τους. Οι σχέσεις πιστωτών οφιλετών είναι κάτι πολύ ευαίσθητο και από πλευράς ανθρωπίνων σχέσεων και είναι πολύ ευαίσθητο ζήτημα στην τσεχική δημοκρατία. Βάσει της εμπειρίας μου γνωρίζω ότι δεν πρέπει να τιμωρεί το κάθε οφειλέτης διότι δεν ήταν αρκετά υπεύθυνο όσον αφορά το χρέος του. Και οι πιστωτές θα πρέπει να διαθέτουν όμως εργαλεία ούτως ώστε με αποτελεσματικό τρόπο να μπορούν να παίρνουν τα χρήματά τους πίσω. Αυτή η έκθεση είναι καλός συμβιβασμός πιστεύω. Αντικατοπτρίζει και, τις, και τα συμφέροντα και των οφειλετών και των δανειστών. Είμαι υπέρ λοιπόν της εκθέσεως και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κοφεράτη, πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, από την αρχή θεωρήσαμε ότι ήταν πολύ σκόπιμη, πολύ θετική, τουλάχιστον όσον αφορά τι προθέσει, η οδηγία που θα ψηφίσουμε αύριο. Πιο συγκεκριμένα, μια στιγμή που οι οικονομικέ και κοινωνικέ συνέπειε τη μακροχρόνια κρίση την οποία διανύουμε δεν έχουν ακόμα αποκατασταθεί. Είναι πολύ καλό να εφαρμόσουμε όλα τα διαθέσιμα νομικά μέσα που θα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να ακολουθήσουν ε, πορείες αναδιάθρωσης που μπορούν να διασώσουν την οικονομική τους δραστηριότητα πρώτα απ' όλα και μετά να βοηθηθούν να ακολουθήσουν τις διάφορες διαδικασίες ε, φερεγγιότητας και έτσι να αποφύγουμε απώλεια θέσεων εργασίας που είναι κάτι που έχει δραματικές κοινωνικές συνέπειες. Το βλέπουμε αυτό συχνά. Το κείμενο θα ψηφίσουμε ένα καρπός μακρών διαπραγματεύσεων που ενδιέφεραν καταρχάς το Κοινοβούλιο και μετά τις συνομιλίες Κοινοβουλίου-Συμβουλίου. Για αυτό το λόγο μπορέσαμε να καλύψουμε πιο ευαίσθητα θέμα, όπως υπενθύμησαν οι προλαλήσαντες συνάδελφοι. Δεν μπορούμε όμως να τη δούμε αρνητικά αυτή την προσέγγιση και την έκθεση, την οδηγία μάλλον. Χάσαμε όμως σημαντική ευκαιρία κατά την άποψή μας να εξασφαλίσουμε καλύτερη προστασία για, τα, για πιο ευάλωτους φορείς σε αυτή τη δραματική φάση που περνάνε Κάποιε ε, περιοχές για αναδιάθρωση επιχειρηματική που εκεί εμπλέκονται πολύ μεγάλες επιχειρήσεις ευρωπαϊκές αλλά πολύ συχνά και περισσότερο μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το σχέδιο αναδιάθρωση δεν αφορά μόνο τα θέματα τα χρηματοπιστωτικά που είναι πιο προφανή ζητήματα σε πολλές περιστάσει και διαφαίνονται αλλά η αναδιάθρωση επεκτείνεται αναπόφευκτα και σε θέματα που άπτονται τη διοργάνωση τη επιχειρήσεω. Όχι μόνο διότι όταν υπάρχουν ελλείψεις δημιουργούνται προβλήματα, αλλά για να φύγουν από τις δυσκολίες επιχειρήσεις πρέπει να αλλάξουν το οργανωτικό τους μοντέλο, που είναι και το αίτιο της ε, κρίσης. Συνεπώς, όσον αφορά την οργάνωση των επιχειρήσεων που των επιχειρήσεων που υποφέρουν, η διαδικασία αφορά επίσης και την αμοιβή των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας. Εννοούμε τον αριθμό των ανθρώπων που εμπλέκονται, με στις συνθήκες συμπεριλαμβάνεται αυτό, και τον ε, τον χαρακτήρα της εταιρείας, της επιχείρησης, τον πολιτιστικό χαρακτήρα επίσης ε, της εταιρείας και των θέσεων εργασίας που μπορεί να απολεστούν. Λοιπόν, θέλαμε να επισημοποιηθεί η ανάγκη μιας συμμετοχής προληπτικής των φορέων και πλήρης ενημέρωσης των εργαζομένων και των άλλων φορέων των εμπλεκομένων όσων έρχονται σε επαφή και συμμετέχουν σε εργασίες της επιχείρησης. Καταφέραμε από αυτή την έποψη ε, να κάνουμε σημαντικά βήματα πρόοδους όπως ε, αναφέρθηκε και γι' αυτό πρέπει να ευχαριστήσουμε και το κάνω πολύ ευχαρίστω την προσπάθεια της συγγήτριας κυρίως κατά τη διάρκεια ενός πολύ μακροχρονίου τριμερούς διαλόγου. Θα έπρεπε όμως να προσθέσουμε και κάποιο άλλο βήμα πρόοδου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προβλέπεται υποχρέωση ε, επιβεβαίωσης εκφράσης της άποψης των εργαζομένων στον αφορά τις αλλαγές στη διοργάνωση επιχείρησης. Ε, ε, προβλέπονται οικονομικέ συνθήκες, ωράρια, απολύσει και διάφορες συνθήκες οι πραγματικές εργασίες. Αυτή η έλλειψη του σημείου για μα είναι μία από τι χαμένε ευκαιρίες για μία καλή νομοθέτηση και μία προόδο όσον αφορά τους πιο αδύναμους φορείς. Ένα άλλο σημείο στο οποίο χάσαμε μία ευκαιρία αφορά και σε αυτή την περίπτωση εργαζομένου. Αυτή τη φορά όχι όμω αν εργατική δύναμη που αφορά και την οργάνωση επιχείρηση, αλλά με τη σειρά του σαν ενδεχόμενοι πιστωτέ μια επιχείρηση που περνάει κρίση. Πιστεύουμε ότι πιστωτέ δεν μπορούν να θεωρούνται όλοι ότι είναι στο ίδιο επίπεδο και θα ήταν χρήσιμο και απαραίτητο να εγγυηθούμε μεγαλύτερη προστασία στου πιστωτέ, που είναι πια δύναμη, του εργαζομένου ακριβώ. Πιο συγκεκριμένα πιστεύουμε ότι η πρόβλεψη ειδική κατηγορία για τις πιστώσει των εργαζομένων πιστωτών δεν θα πρέπει να επαφίεται στην κρίση των κρατών μελών, θα έπρεπε να είναι κάτι υποχρεωτικό. Θα ήταν επίση ενδεδειγμένο σε αυτή την τάξη να δίνονται προτιμησιακέ προσεγγίσει και πρόσθετε προστασίε εν συγκρίση με τι άλλε κατηγορίε πιστωτών. Σταματάμε εδώ. Είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό. Αλλά θέλουμε αύριο όμως να εγκριθεί αυτή η οδηγία. Αλλά προβλέπω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε την επεξεργασία μέχρι ότου αυτή Αυτές οι ευκαιρίες που χαθήκαν μέχρι τώρα, τελικά στο μέλλον, κυρίως για το νέο κοινοβούλιο που θα εκλεγεί από τους Ευρωπαίους πολίτες τις επόμενες εβδομάδες, να είναι ευκαιρία στο νέο κοινοβούλιο να επανέλθει επί του θέματος και να εγγυηθεί αποτελεσματική πρόοδο εποφελή για όλους, και για την επιχείρηση και για το εργατικό δυναμικό. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ένα λεπτό. Σόσνιας. Ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε, αλλά δεν καταλαβαίνω. Πού θα τα βρείτε τα λεφτά αυτά για να σώσετε όλες αυτές τις αποτυχημένες επιχειρήσεις. Από τα περντίεμ που παίρνετε κύριοι ευρωβουλευτές ή από την τσέπη των φορολογουμένων. Α, και άλλα λεφτά που θα πάνε από τις ε, καλές επιχειρήσει που πληρώνουν φόρο, τι βιώσιμε, θα πηγαίνουν ε, στις αποτυχημένε, στι φαληρημένες. Αυτού που χάνουν δηλαδή στο παιχνίδι του ανταγωνισμού. Για να σώσουμε ίσως ε, μία θέση εργασία σε μία αναποτελεσματική εταιρεία θα θυσιάσετε δύο θέσει εργασία σε μία επιτυχημένη εταιρεία. Και επίση θα πληρώσουμε και για τους υπαλλήλους οι οποίοι θα ασχοληθούν με την περίπτωση Μα τι πράγματα είναι αυτά. Δεν είναι πολύ σωστή αντιμετώπιση. Δεν είναι σωστή χρήση αυτή των δημοσίων πόρων. Στην ουσία δίνετε χρήματα, κάνετε αναδιανομή. Ε, χρήματα από τους μεν δε μέσω διοικητικών μεθόδων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ράντεφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Συγχαίρω την κυρία Νίμπλερ για τη συμφωνία επί της οδηγίας για τι προληπτικέ ε, αναδιαρθρώσει, ε, τη δεύτερη ευκαιρία και τα μέτρα για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των ε, αναδιαρθρώσεων, αφαιρεγιωτήτων και τη διαδικασία απαλλαγή. Είναι πολύ γνωστό ότι οι αποτελεσματικέ διαδικασίε σε περιπτώσει αφαιρεγιότητα είναι πολύ καλέ για το επιχειρηματικό κλίμα, βοηθούν τη δημιουργία θέσεων εργασία, αποτρέπουν απόλυτα θέσεων εργασία και βοηθούν να αντιμετωπίσουμε τι κυκλικέ υφέσει και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των μη εξυπηρετημένων δανείων και τη ανεργία. Οι διαφορές μεταξύ των εθνικών διαδικασιών μπορούν να κάνουν τη διαδικασία προστασία των συμφερόντων των εταιριών ιδιαίτερα μακροχρόνιε. Αυτό ε, δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία τη αγορά και των εθνικών οικονομιών. Η αβεβαιότητα είναι αποτρεπτικός παράγοντας για διαμεθοριακές επενδύσεις. 1,7 εκατομμύρια εργαζόμενοι χάνουν κάθε χρόνο την εργασία τους λόγω πτωχεύσεων. Έτσι θα βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υποφεληθούν από αυτή τη δεύτερη ευκαιρία και από τα βασικά, ε, τις βασικές αρχές της ε, προληπτικής αναδιάρθρωσης και από απλούστερη διαδικασία αφαιρεγγιότητας. Έτσι θα μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα στις υποχρεώσεις τους και θα σταματήσει αυτή η διαδικασία μονίμων οφειλετών. Θα μειωθεί η έκθεση των τραπεζών σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια και θα αντιμετωπιστεί συσσόρευση τέτοιων, δανείων, τέτοιων κακών δανείων στο μέλλον. Αυτό πρέπει να ισχύσει όμω και στου καταναλωτέ. Γι' αυτό πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη θα λάβουν υπόψη τι συστάσει που γίνονται και θα αρχίσουν να αντιμετωπίζουν την υπερχρέωση εισάγοντας υποχρεωτικούς ε, κανόνες για τις απαλλαγές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ράτεφ. Δεν έχει ζητήσει κανείς άλλος. Α, κύριε Ράτεφ, επιτρέπετε γαλάζια κάρτα από τον συνάδελφο Σόσνιτς. Δέχεστε μια ερώτηση από τον συνάδελφο Σόσνιτς. Πείτε. Παρακαλώ. Η ερώτησή μου είναι εξής. Πώς θέλετε να αυξήσετε ε, τη ε, δανειοληπτική ε, ικανότητα των εταιριών. Το χρήμα για να κυκλοφορεί πρέπει να ρέει προς τη μία την άλλη κατεύθυνση. Οι τράπεζες ενθαρρύνουν τις εταιρείες να αναλαμβάνουν μεγαλύτερους κινδύνους, άρα να είναι και στο χείλος της χρεοκοπίας. Όταν υπάρχει μια τέτοια διαδικασία ε, με σαφείς κανόνες προκαθορισμένους, τότε ε, μπορεί ε, αυτό να βοηθήσει ακόμα και στη μερική απαλλαγή και μπορεί να μείνει βιώσιμη μια μικρομεσαία επιχείρηση και να μην κάνει απολύσεις. Αυτό είναι προς όφελος και των δανειοληπτών και των τραπεζών και της σύνολης οικονομίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ράντεφ. Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το λόγο τώρα έχει ο Επίτροπος κύριος Κίνγκ. Um, Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση και ευχαριστώ όλου για τη ε, δουλειά που κάνατε για αυτό το ντοσιέ και το σημείο στο οποίο φτάσαμε. Εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλω απλώ να σα ενθαρρύνω να υπερψηφίσετε την πολιτική συμφωνία για την οδηγία για την αφαιρεγκαιότητα που επετέχθη τον Δεκέμβριο σε ό,τι αφορά τη δική μα την πλευρά θα εργαστούμε άοκνα για να βεβαιωθούμε ότι όταν το Συμβούλιο ολοκληρώσει τι σχετικέ διαδικασίε, η οδηγία τάχιστα και αποτελεσματικά θα μεταφερθεί και θα υλοποιηθεί από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, κύριε Κίνγκ. Για να κλείσει η συζήτηση, το λόγο έχει η συγγήτρια κυρία Νίβλε. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχά θέλω να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Επιτροπή Κίνγκ, αλλά και τους συναδέλφους οι οποίοι εργάστηκαν σε αυτό το θέμα με μεγάλο ενθουσιασμό. Θέλω να τονίσω και πάλι ότι πιστεύω πως φτάσαμε σε ένα πάρα πολύ καλό συμβιβασμό που θα προωθήσει την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη και έτσι κάναμε ένα σημαντικό βήμα πρόοδου σε όλα τα κράτη-μέλη έχουμε τόσους πολλούς ταλαντούχους ανθρώπους, τόσα γερά μυαλά. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε και τους νέους να αναλαμβάνουν τον κίνδυνο, να ιδρύουν μια επιχείρηση και εκεί οδηγεί συγκεκριμένη οδηγία, η οποία σε περίπτωση δυσχεριών ε, θα τους βοηθήσει να αναδιαρθρώνονται ή να αποκτούν μια δεύτερη ευκαιρία. Τώρα ο συνάδελφος που είπε ότι εδώ, εδώ έχουμε κάνει αυτό για να κυκλοφορούν λεφτά σε διάφορες κατευθύνσεις, αυτά είναι ανοησίες. Δεν είναι κρατικές ενισχύσεις αυτές. Είτε θα αφήνουμε τις εταιρείε να πτωχεύουν, είτε θα βρούμε ένα ευφύ τρόπο να τις βοηθούμε με μεταφορά του χρέους για να υποστηρίζεται μια ε, εταιρεία που μπορεί συγκυριακά να έχει κάποιες δυσκολίες και να θέλει μια βοήθεια σε αυτό εξυπηρετεί συγκεκριμένη οδηγία λοιπόν και χαίρομαι που προχωρήσαμε τόσο πολύ χωρίς να ε, αποδυναμώνουμε κανέναν. Θέλουμε να ενισχύσουμε τις εταιρείε. Δεν ζητάμε απλώ κρατικές ενισχύσεις, χρειαζόμαστε τις εταιρείε που να επενδύουν, που να αναλαμβάνουν κίνδυνο και να δημιουργούν θέσεις εργασίας. Ακριβώς αυτές πρέπει να βοηθούμε και να το κάνουμε ε, κάναμε τη δουλειά μας. Ελπίζω αύριο να γίνει δεκτή η έκθεση με μεγάλη πλειοψηφία και πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία ε, για να ενισχύσουμε και τους εργαζομένους. Κύριε Κοφεράτη, στο παρελθόν πάντα είχαμε τη συζήτηση ε, χρειάζονται καλύτερη υποστήριξη, όχι απασχολούμενοι. Πάντως, σε πολλές συζητήσεις που είχαμε και ενημερωτικές και διαπραγμάτευσης, ε, καταλήξαμε, δεν δεχτήκαμε προτιμησιακά δικαιώματα. Έχουν τα δικαιώματα εργαζομένοι τα ίδια με εκείνα που έχουν όλοι οι υπόλοιποι πιστωτέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. εγώ ευχαριστώ κύριε Νίβλερ. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο, όπω είπε η συγγήτρια. Επόμενο θέμα στην μέση διάταξη, έκθεση του κυρίου Σβόμποτα άσκηση των δικαιωμάτων πραγματικής ιδιοκτησία και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταθώσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων. Για τέσσερα λεπτά έχει το λόγο ο εισηγητής κύριε Φόμποντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που θα ψηφίσουμε για το αποτέλεσμα τη διαπραγματεύση, μια διαπραγμάτευση που δεν ήταν καθόλου εύκολη. Θέλω να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου και όλου του εκπροσώπου των υπολείπων θεσμικών οργάνων για την υπομονή του και για την αποφασιστικότητά του να καταλήξουμε σε συμφωνία. Ιδιαίτερα τη συνάδελφο κυρία Νίμπλερ. Η εφαρμογή τη ενιαίας ψηφιακή ε, αγορά είναι προτεραιότητα τη Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η θέση του Κοινοβουλίου διέφερε από αυτήν της Κομισιόν. Οπότε ήταν υποχρέωσή μας να δράσουμε σύμφωνα με τη γνώμη της πλειοψηφίας των συναδέλφων. Πιο συγκεκριμένα το, το Κοινοβούλιο θεωρούσε ότι θα έπρεπε να στηρίξουμε τους δημιουργούς και να τους χορηγήσουμε μια νομική ασφάλεια στα μακρόπνοα σχέδιά τους. Πάντα λέγαμε ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε την πολυμορφία της ευρωπαϊκής, ε, του ευρωπαϊκού πολιτιστικού προϊόντος και να παράσχουμε τις κατάλληλες συνθήκες ε, στους ε, Ευρωπαίους δημιουργούς. Να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για τις μεταδόσεις και αναμεταδόσεις προγραμμάτων. Ταυτόχρονα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και ένα ασφαλές περιβάλλον για τις ε, ψηφιακές ε, επιχειρήσεις. Γι' αυτό το λόγο εφαρμόσαμε την αρχή της ε, χώρας προέλευσης. ο συμβιβασμός στον οποίο καταλήξαμε είναι ισορροπημένος και θα επιτρέψει στα, στους ε, ραδιοτηλεοπτικούς ε, φορείς να μεταδίδουν προγράμματα ε, επιγραμμικά στο ίντερνετ και να τα πολλούν. Οι κατανοητέ από την άλλη μεριά θα έχουν μεγαλύτερη ποικιλία προγραμμάτων που μπορούν να παρακολουθήσουν από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Το Κοινοβούλιο επίσης ζήτησε να διασφαλιστεί ο ε, η δυνατότητα της άμεσης προσφυγής κάτι που σημαίνει ότι ο κανονισμός θα έπρεπε να γίνει να μετατραπεί σε οδηγία. Αντιμετωπίσαμε αυτή την αλλαγή και θα ψηφίσουμε για μια οδηγία, όχι για ένα κανονισμό. Η εφαρμογή των κανόνων θα διέπεται από την ε, επιθυμία να εξασφαλίσουμε τα πνευματικά δικαιώματα, το copyright και να προσπιστούσουμε τα δικαιώματα τόσο των παραγωγών, των δημιουργών, όσο και των καταναλωτών. Νομίζω ότι η συμφωνία είναι ένας ισορροπημένος συμβασμός και ε, επιφυλασσόμεθα να, λάβουμε περισσότερα, να κάνουμε περισσότερα βήματα αν αλλάξει η σημερινή κατάσταση. Καλό λοιπόν τους συναδέλφους να στηρίξουν αυτό το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σφόποτα. Για τρία λεπτά η κυρία Γουόρτ παρακαλώ. I welcome. Καλωσορίζω την απόφαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκολύνει τη διαθεσιμότητα των πολιτιστικών αγαθών σε όλα τα κράτη-μέλη. Είναι σημαντικό οι επιγραμμικές υπηρεσίες ε, να καλλιεργούνται, αλλά να μην έχουμε και φραγμούς διασυνοριακά, ενώ προστατεύουμε τα συμβεσιακά δικαιώματα των παραγωγών και των υπεύθυνων για τι ρεπετελεοπτικέ εκπομπέ. Είναι σημαντικό για τον πολιτιστικό τομέα να παραμένει ένα ικανοποιητικό επίπεδο ελέγχου στο, ε, σε ό,τι παράγουν. Ε, η νομοθεσία αυτή προβλέπει κάποια βήματα πρόοδου για του καταναλωτέ και θα αυξήσει τη, διαθεσιμότητα κάποιων ε, προγραμμάτων σε όλη την Ευρώπη και εκπομπών. Ε, αυτό είναι σημαντικό και για του παραγωγού και για του πολίτε που έχουν σχέση με τα πολιτιστικά. Η ενημέρωση και οι καθημερινέ ειδήσει θα είναι πιο εύκολα προσβάσιμε. Έτσι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικέ ειδήσει και μέσα μαζική ενημέρωση οι πολίτε σε όλη την Ήπειρο. Και αυτό θα έχει μια πολύ καλή ευεργετική συνέπεια για όλους. Ε, διότι μπορούμε να προβλέψουμε καλύτερη ποιότητα εκπομπών σε όλη την Ευρώπη. Ελπίζω λοιπόν να ε, αναπτύξουμε έτσι μια καλύτερη ευρωπαϊκή προοπτική κοινή για τις καθημερινές εξελίξεις. Θα πρέπει για τις εκπομπές αυτές να δούμε ότι η αρχή είναι, ε, της χώρας προέλευσης είναι καλή ιδέα γιατί αυξάνεται η δυνατότητα πρόσβασης όλων. Θα επιτρέψει ο κανονισμός αυτός στις προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης να προβλέψουν για διθεσιμότητα των πολιτιστικών αγαθών, ενώ θα προστατεύονται και συμπεσιακέ ελευθερίε. Ο πολιτισμό και η κουλτούρα είναι σημαντική για την δημιουργία ισχυρών δεσμών μεταξύ των χωρών τη Υπήρου και για να καταλύει του φραγμού μεταξύ των ανθρώπων. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε τον πολιτισμό ως μια κοινή εμπειρία που διαμορφώνεται για όλου μα ταυτόχρονα. Ένα υγιή τομέα ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών που φτάνει σε όλου του πολίτε παντού είναι σημαντικό πυλώνα. Με αυτό το νομοθέτημα θα πρέπει να σκεφτούμε και τους πνευματικούς δημιουργούς και τους παραγωγούς. Όσοι δημιουργούν το περιεχόμενο δεν πρέπει να είναι ευάλωτοι στην εκμετάλλευση και να λαμβάνουν ή, ε, την, την αμοιβή που αξίζουν για την παραγωγή τους. Θα πρέπει οι κάτοχοι πνευματικών ε, δικαιωμάτων να προστατεύονται από τον νόμο ώστε να έχουν δίκαιη ανταμοιβή. Ποτέ δεν πρέπει αυτοί που κάνουν τις εκπομπές να υποφελούνται δυσανάλογα από τη δουλειά άλλων. Η προστασία των ε, ε, όσων παράγουν τα πολιτιστικά αγαθά έχουν να κάνουν ακριβώς με την προστασία του ίδιου του τομέα. Θα πρέπει το εισόδημά τους να είναι εγγυημένο, θα πρέπει να μπορούν να διοπορίζονται. Ιδάλλως μπορεί να καταστρέψουμε την όλη ποικιλομορφία του τομέα αυτού. Θα ήθελα λοιπόν να ρίξουμε μια ματιά και προς το μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι θα συνεχίσουν να μειώνονται οι φραγμοί στις διαδικτυλοπτικές εκπομπές ε, όλη την Ευρώπη. Αυτό διαρκώ θα βελτιώνει την ποιότητα των προγραμμάτων και εκπομπών που διατίθενται. Ωστόσο, δεν μπορούμε απλώ να διευκολύνουμε τα βελτιωμένα προγράμματα χωρί να προσφέρουμε στήριξη σε ανεξάρτητου και εναλλακτικού και εναλλακτικούς φορεί που παράγουν τηλεοπτικό υλικό. Θα πρέπει σε όλου σε όλη την Ευρώπη να προσφέρουμε το ίδιο δίκτυο Προστασία και να μην επιτρέπουν στην Ευρώπη να δεσπόζουν μικρέ οργανώσει που συγκεντρώνουν πολλά στα χέρια του από μικρέ περιοχέ. Ευχαριστώ κύριε Γόρτα, εξ ονόματος τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το λόγο έχει ο Επίτροπο κύριος Κίνγκ. Χαίρομαι που συζητάμε την πολιτική συμφωνία στην οποία καταλήξαμε για αυτή την πρόταση. Εκ μέρου τη Κομισιόν συμφωνήσαμε, συμφωνούμε ότι αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό κομμάτι της ε, Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Στρατηγικής. Εκ μέρους των συναδέλφων θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συζητητές και όλους όσοι συνεισέφεραν. Η οδηγία θα μας επιτρέψει να ωφεληθούμε περισσότερο από την πολιστική ε, ποικιλία ε, καθιστώντας πιο εύκολη την απόδοση του copyright των δικαιωμάτων των πνευματικής ιδιοκτησίας σε, ε, σε ραδιοτηλεοπτικούς φορείς. Επίσης, ε, θα ε, βοηθήσουμε τις διάφορες γλωσσικές μειονότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν προγράμματα στη γλώσσα τους. Με ε, συγκεκριμένα μέτρα προστασίας. Η τηλεο, ραδιοτηλεοπτικοί φορείς πλέον μπορούν να ε, εμπορεύονται το περιεχόμενό τους μέσω του ίντερνετ, να, έχουν, να παίρνουν δικαιώματα τέτοια συμμετάδοση ή αναμετάδοση σε άλλα κράτη-μέλη και περιλαμβάνονται επίσης και κανόνες για την ε, τεχνική που, της, ε, ε που θα χρησιμοποιηθεί για την ανταπόδοση, την αμοιβή των δημιουργών. Δυστυχώ, η αρχική νομική βάση βέβαια που προτάθηκε το άρθρο 114 αντικαταστήθηκε με τα άρθρα 53, 1 και 62. Ε, σκοπεύουμε να υποβάλουμε μια συγκεκριμένη δήλωση από την Κομισιόν για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Για να κλείσει η συζήτηση, το λόγο έχει ο Σόβοντα και πάλι εισηγητής για δύο λεπτά. Um Ζητώ συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. Ε, όλα λάθος τα είπα. Ε, δεν βλέπω τον κύριο Μπούζεκ. Γι' αυτό το λόγο έχει η κυρία Μπουτονέ τώρα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχά θα ήθελα να ευχαριστήσω του συναδέλφου ιδιαίτερα την κυρία Νίμπλερ, για την εξαιρετική της εργασία στην Επιτροπή και στις διοργανικέ διαπραγματεύσεις. Το κείμενο που θα ψηφίσουμε αύριο ε, θα εξασφαλίσει ίση πρόσβαση παντού στην Ευρώπη για άλλους πολίτες και ε, θα διευκολύνει την ίσπραξη πνευματικών δικαιωμάτων από τους ε, ε, λόγω φορείς. Η ε, ε, πρόταση κανονισμού έγινε πρόταση οδηγία, αφήνοντα έτσι κάποια διακριτική ευχαίρεια στα κράτη-μέλη. Η εφαρμογή της αρχής της χώρας προέλευσης περιορίζεται στις ενημερωτικές εκπομπές, στις ειδήσει και στις εσωτερικές παραγωγές που χρηματοδοτεί 100% ένας ραδιοτηλεπτικός οργανισμός. Ε, παραμένει αρχή ε, η εντοπιότητα ε, και έτσι διαφυλάσσεται η ποικιλομορφία πολιτιστική και γλωσσική. Και τέλος, ε, με την ε, άμεση μετάδοση απευθείας διευκρινίζεται η κατάσταση και διευκολύνεται. Έτσι οι δικαιούχοι των δικαιωμάτων θα έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου. Η πρόταση οδηγίας αυτή είναι σημαντική για τους πολίτες μας, τους ε, δικαιούχους των δικαιωμάτων και τη διαφύλαξη μιας ποιοτική πολιτισμικής προσφοράς. Ευχαριστώ κυρία Βουτονέ. Τώρα ακολουθεί η διαδικασία Η κυρία Νίμπλερ ζήτησε το λόγο στο Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά τον εισηγητή μας και πρόεδρο της Επιτροπής ε, που σε πάρα πολλούς ε, τριμερείς διαλόγους ε, μας βοήθησε με την πραγματογνωμοσύνη του και με την ηγεσία του. Χωρί τον κύριο Σβόμποντα δεν θα είχαμε προχωρήσει. Κυρίω γι' αυτό ζήτησα το λόγο εγώ για να επενέσω τον εισηγητή, αλλά και οδηγία είναι ορόσημο διευκολύνουμε τη διάδοση στο διαδίκτυο, τη μετάδοση και αναμετάδοση, ε, την χορήγηση των πνευματικών δικαιωμάτων. Παντού θα είναι πιο εύκολη η πρόσβαση, αλλά με δίκαιες προϋποθέσεις και όρους. Και αυτό είναι σημαντικό για μένα. Βρήκαμε λοιπόν μια σωστή ισορροπία ανάμεσα ε, στην ε, προστασία εκείνων που δημιουργούν ταινίε και τα συμφέροντα των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών. Οι συμπαραγωγές επίσης θεωρώ ε, πραγματικά να τονίσω ότι εξαιρούνται ε, και ε, για να μπορούν να χρηματοδοτούνται οι ταινίε. Η Ευρώπη δεν είναι μόνο μια αγορά, αλλά ζει από την ποικιλομορφία των πολιτισμών της. Και ελπίζω να μπορέσουν όλοι οι Ευρωπαίοι να επωφεληθούν. Ο πρόεδρο διακόπτει την ομιλήτρια και τη αφαιρεί το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Νίβλερ. Δικασία Κατσιά ολοκληρώθηκε εδώ και πάλι ο Επίτροπο κύριο Κίνγκ εξ ονόματο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, η σημερινή συζήτηση είναι πάρα πολύ σύντομη. Ελπίζω αυτό να μην δείχνει ότι το θέμα δεν έχει σημασία. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πρόταση. Θα συνεισφέρει έτσι ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση σε περιεχόμενο, ραδιοτηλεοπτικό περιεχόμενο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου στην ολοκλήρωση τη ενιαία ψηφιακής αγοράς της Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν, δεν είναι κάτι θεωρητικό. Θα αλλάξει τα πράγματα στην πράξη, θα δώσει μεγαλύτερη πρόσβαση σε ραδιοτηλεοπτικό περιεχόμενο ε, διαμέσου των συνόρων. Κατά την άποψή μα, θα πρέπει να γίνει πραγματικότητα το συντομότερο δυνατό και θα παρακολουθήσουμε την εφαρμογή αυτή τη οδηγία. Ε, ελπίζω ότι θα υπερψηφιστεί αύριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πίτροπε, κύριε Κίνγκ. Λοιπόν, τώρα έχει το λόγο η συγκητή για να κλείσει η συζήτηση. Παρακαλώ, κύριε Σπαπούτα. Πρόεδρε, Επίτροπε, eh, eh, eh, η συζήτηση δεν δείχνει να υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες σε ό,τι φορά αυτή την πρόταση. Και χαίρομαι ιδιαίτερος που αύριο μπορούμε να ελπίζουμε ότι αυτό το βήμα προς την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς θα υπερψηφιστεί. Ελπίζω ότι οι προσδοκίες ε, της Επιτροπής ε, στην αρχή αυτής της διαδικασίας ήταν κάπως υψηλότερες από το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. παρόλα αυτά ε, θα προχωρήσει. Το 1950 ο Σούμαν είπε ότι την Ευρώπη δεν μπορούμε να την κάνουμε με πολλά βήματα διαδοχικά. Αυτό ισχύει λοιπόν και για αυτή την πρόταση. Θα πρέπει να περιμένουμε και βαθμιδών να δημιουργήσουμε τα υπόλοιπα που χρειάζονται. Ε, η νομοθεσία λοιπόν αυτή θα μπορεί να επεκταθεί και να διευρυνθεί το πεδίο της. Ελπίζω ότι η θαυμάσια συνεργασία που είχαμε με την Επιτροπή και την κυρία Νίμπλερ θα είναι ε, ιονό και για μελλοντικέ ε, ανάλογε διαπραγματεύσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σπόποτα. Ολοκληρώνω τη συζήτηση εδώ λοιπόν. Ε, τελευταίο θέμα για απόψε είναι η συζήτηση της έκθεσης Βάουτμανς, απόφαση για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη. Το λόγο έχει για πέντε λεπτά η συγγήτρια. Κυρία Βάουτμανς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, ε, συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Αύριο θα ψηφίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια σημαντική σύσταση. Μια σύσταση για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη. Ένα νέο ταμείο ε, εκτός προϋπολογισμού 10,5 ε, δισεκατομμύρια για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Είναι ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο που θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, προχωρήσει σε ε, δραστηριότητες και στρατιωτικές και αμυντικές ε, πιο ευέλικτα. Πώς θα γίνει αυτό. Είχαμε διάφορα μέσα για την εξωτερική πολιτική τα οποία συγκεντρώνουμε κάτω από μία ομπρέλα χρηματοδοτική για να καλυφθούν πολλά κενά που υπάρχουν και ελλείμματα. και έτσι θα μπορούν να χρηματοδοτούνται ε, πιο εύκολα κάποιες δράσεις γιατί στο παρελθόν υπήρχε προϋπόθεση αναπτυξιακής βοήθεια και δεν μπορούσαμε να υποστηρίζουμε κάποιες ειρηνευτικές δράσεις, ιδιαίτερα στην Αφρική. Ε, τώρα υπάρχει αυτός ο μηχανισμός για την ειρήνη ε, και θα αλλάξει όλη την κατάσταση. Πρώτα, θα φροντίσουμε να υπάρχει μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών με καλύτερο επιμερισμό των βαρών. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός ε, για την Ειρήνη θα έρθει να αντικαταστήσει το μηχανισμό Αθήνα. Ε, μέχρι 45% θα είναι χρηματοδότηση. Βεβαίω, τα κράτη-μέλη ε, πιο εύκολα θα τείνουν να συμμετέχουν σε δράσεις και επιχειρήσεις. εάν είναι περισσότερο το κοινοτικό κόστος, έχει λιγότερο κόστος το κάθε κράτος μέλος να υπομειστεί. Δεύτερον, μπορούμε να υποστηρίζουμε ερνευτικέ επιχειρήσει των διεθνών οργανισμών και τρίτων χωρών και δεν θα περιοριζόμαστε μόνο στην Αφρική, μπορούμε να έχουμε και ένα ευρύτερο πεδίο. Και το τρίτο και σημαντικό επίση θα μπορέσουμε να συνεισφέρουμε ε, σε ικανότητες στρατιωτικές και αμυντικές τρίτων χωρών. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Στη Σομαλία έχουμε εκπαιδευτικές αποστολές, όπου μπορούμε εμείς να εκπαιδεύσουμε ε, τους ε, ε, στρατιώτες εκεί. Αν δεν έχουμε όμως το υλικό, αν δεν έχουμε αλεξίσφαιρα γυλαίκα, τι να την κάνουν την εκπαίδευσή μας. Έτσι θα διευκολύνεται και η παροχή βοήθειας. Υπάρχει και ρήτρα ευελιξίας. Ε, για να μπορούμε στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας να χρηματοδοτούμε ε, τέτοιες δράσεις. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Ειρήνη είναι ένα ταμείο εκτός του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Για μένα αυτό τι σημαίνει ότι ε, θα πρέπει το κοινοβούλιο μας να έχει και λόγο και κοινοβουλευτικό έλεγχο στο ταμείο αυτό. Θα πρέπει ε, εν γέρος να ενημερωνόμαστε και να λαμβάνουμε υπόψη την κατάσταση για να αποφαινόμαστε και να εξασφαλίζουμε ότι δεν θα χρηματοδοτούνται δράσεις που αντιβαίνουν στο άρθρο 21 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το μέσο αυτό θα είναι συμπληρωματικό με άλλα μέσα άσκηση εξωτερικής πολιτικής. Κύριε Πίτροπε. Πολύ συχνά διαμαρτυρόμαστε και γκρινιάζουμε και ακούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε θέση να δρά ή δρά πολύ καθυστερημένα ή ε, δρά χωρίς θένος. Ε, τώρα ε, ο κόσμος μας είναι πολύ πιο περίπλοκος, πολύ πιο απρόβλεπτος, πολύ πιο επικίνδυνος και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαθέτει νέα μέσα για να προλαμβάνει σειράξεις και να εξασφαλίζει τη διεθνή ασφάλεια και βεβαίως να παίζει και το ρόλο της ε, ως παγκόσμιος πρωταγωνιστής ε, στην ασφάλεια και στην ειρήνη. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Ειρήνη, συνάδελφε, είναι πραγματικά εδώ αναπόσπαστος κρίκος σε αυτή την προσπάθεια. Και σας παρακαλώ να εγκρίνετε τη σύσταση αυτή ε, με μεγάλη ενέργεια και χαρά. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Ελπίζω αύριο να ε, βρει μια μεγάλη πλειοψηφία η σύσταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Βότμαν. Σε ξενόμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Κίνγκ. Ε, ε. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όλοι σας ξεχωριστά. Εκ μέρου τη είπα τη εκπροσώπου, να σα ευχαριστήσω για την ευρεία στήριξή σα, για την πρόταση να δημιουργήσουμε τη διευκόλυνση για την ειρήνη. Αυτό αντικατοπτρίζει την ανάγκη που επανειλημμένω έχει τονίσει και το σώμα σα να έχουμε χρηματοδότηση στον τομέα αυτό που να είναι πιο ευέλικτη και αποτελεσματική, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη αλληλεγγύη. Επιτρέψτε μου, εκ μέρου τη ΥΠΑ τη εκπροσώπου και των υπόλοιπων συναδέλφων, να επαναλάβω ευχαριστίε προ την εισηγήτρια την κυρία Βότμαν και του συνεισηγητέ τη ε, για την αφοσίωσή του προ το σκοπό τη δημιουργία μια πραγματιστική προσέγγιση. Ε, ε, ε Όπω τονίζετε και εσεί στην έκθεσή σα, ο σκοπό τη Ένωση είναι να είναι πρωταγωνιστή στο διεθνέ προσκήνιο. Και αυτό είναι μέρο των στρατηγικών μα συμφερόντων. Η εικόνα των απειλών που παρουσιάζεται μπροστά μας μας αναγκάζει να έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε σε μια σειρά απειλών κατά της ασφαλείας μας. Αυτό αναφέρθηκε και στα πλαίσια της σφαιρικής στρατηγικής της Global Strategy του 2016 και θα πρέπει να βασιστούμε στις κοινέ μας εμπειρίες όπως τόνισε και ο εισηγητής. Η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, δραστήρια στα πράγματα όταν χρειάζεται, όμως πρέπει να δούμε και τι περισσότερο μπορούμε να πετύχουμε. Είχαμε δυσκολίες να χρηματοδοτήσουμε την ε, εκπαίδευση στρατιωτών στη Σομαλία για την κεντροαφρικανική δημοκρατία. Έπρεπε να προσφέρουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό για να συμπληρώσουμε την ε, μετάβασή τη από τον εμφύλιο πόλεμο σε μια σύγχρονη εύρυθμη δημοκρατία. Οι στρατιωτικέ επιχειρήσει πολλέ φορέ ε, πιέζουν πολύ τι χώρε που πρέπει να προσφέρουν στρατεύματα ε, και όχι το ίδιο αυτούς που ασχολούνται με την συμμετοχή και την ανάπτυξη των δυνάμεων. Θα πρέπει λοιπόν στο Συμβούλιο να δούμε πώ μπορεί να ε, αλλάξει κάτι, ώστε η Ένωση να έχει πλέον τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί όλε τι επιχειρησιακέ τη δράσει στα πλαίσια τη κοινή πολιτική άμυνα και ασφάλεια και με τα απαραίτητα στρατιωτικά μέσα για να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα στι ανάγκε. Συγκεκριμένα υπάρχουν τρει βασικέ κατευθύνσει που μπορεί να ε, προωθήσει η ε, διευκόλυνση για την ειρήνη. Πρώτα απ' όλα θα καλύπτει το κοινό κόστο των στρατιωτικών επιχειρήσεων και αποστολών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μεγαλύτερο κόστο θα πρέπει να, να χρηματοδοτείται από κοινού και έτσι θα καλύπτεται καλύτερα και τι ε, επιχειρησιακέ μα ανάγκε και θα ε, βελτιώνεται η ανάπτυξη των ε, στρατιωτών. Επίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμβάλλει στι στρατιωτικέ ειρηνευτικέ αποστολέ σε συνεργασία με άλλου διεθνεί φορεί. Και τρίτον, θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει τι ένοπλε δυνάμει χωρών με τι οποίε συνεργαζόμαστε στα πλαίσια τη στρατιωτική αλλαγή και συνδρομή, όταν αποφασίσει έτσι το Συμβούλιο. Θα πρέπει επίση οι δράσει αυτέ να ορίζονται στο πεδίο τους ε, από το ίδιο το Συμβούλιο. Είναι σαφές ότι κάθε στήριξη προς τους εταίρους μας θα υπόκειται σε αυστηρότατα κριτήρια και ελέγχους, όπως το σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Επίσης, ε, είπα πρόσωπος, προτείνει κάτι το οποίο όλη η Επιτροπή υποστηρίζει βάσει του άρθρου 31 και ε, ο σκοπός είναι να βοηθήσουμε ή να καλλιεργήσουμε σχέσεις συνεργασίας με άλλα οικονομικά ε, εργαλεία που διαθέτουμε, μηχανισμούς χρηματοδότησης, με την ε, χρηστή οικονομική διαχείριση ως ακρογωνιαίο λίθο. Πρόεδρε, να τονίσω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα της κοινή μας προσπάθειας, ώστε να γίνει η πυρός μας πιο ασφαλής, να στηρίξουμε καλύτερα τους εταίρους μας ανά τον κόσμο και να βοηθήσουμε να διαφυλαχθεί το πολυτιμότερο κοινό μας αγαθό, η ασφάλεια κυρία σας Σα ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για την υποστήριξή σα για αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία και ανυπομονώ για τη συζήτησή μα και την υπερψήφιση τη πρόταση αύριο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πέτροπε. Κύριε Κέγκ, για δυόμιση λεπτά ο κύριος Μπένι Φέι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, η υποστήριξη για την ε, ε με διευκόλυνση για την ειρήνη βασίζεται στη στενή συνεργασία των κρατών μελών στα πλαίσια τη κοινή πολιτική άμυνα και ασφάλεια. Είναι μηχανισμό εξορθολογισμού των υπαρχόντων μηχανισμών. Ω ε, Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεισφέρουμε στην πρόταση τη ύπαρξη τη εκπροσώπου όσο περισσότερο μπορούμε. Είναι σαφή ε, η αίτηση οι στατιωτικέ μα δυνατότητε να συνδυαστούν με ένα συνεκτικό μέσο και βάσει τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και του Διεθνού Δικαίου. Επίση, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει αυστηρό έλεγχο από την πλευρά του ίδιου του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο διαρκώ να ενημερώνεται για την ε, πρόσβαση ε, στα χρηματοδοτικά μα μέσα από τι στατιωτικέ επιχειρήσει. Το ίδιο και για τον εξοπλισμό που θα αποστέλλεται ενδεχομένω και στα τρίτα κράτη. Θα πρέπει να συνάδει με την θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την εξαγωγή όπλων και το καθεστώ ε, τη χρήση όπλων, τη διπλή χρήση όπλων. Θα πρέπει επίση να υπάρχει λεπτομερής καταγραφή των εξοπλισμών που παρέχεται. Είναι απαραίτητη η ασφαλιστική, ε, ασφαλιστική δικλίδα αυτή, διότι δεν μπορεί να είναι η στρατιωτική συνεργασία πιο σημαντική από την ειρήνη και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι στα θεμέλια του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο που στο κείμενο προβλέπεται μια πρόταση για τη μνήμα στην μη εξάπλωση και τον αφοπλισμό και ε, στην καταπολέμηση τη ε, ε, διάδοση των πυρηνικών όπλων στην Ευρώπη. Θα πρέπει και η κοινωνία των πολιτών να αναλάβει τι ευθύνε τη και να σταματήσει να πιστεύει ο πολιτικό κόσμο ότι είναι φάσμα του παρελθόντο τα πυρηνικά όπλα. Θα πρέπει να ακούσουμε τα αιτήματα των Ευρωπαίων πολιτών και να σεβαστούμε και τι αρχέ του διεθνού δικαίου που επιτρέπουν στην Ευρώπη να γίνει πρωταγωνίστρια Ευχαριστώ για ένα λεπτό, κύριο Πιμέντα Ευχαριστώ, Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Ειρήνη προτείνει η Κομισιόν. Είναι ένα ακόμα παράδειγμα του πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταφύγει τις πολιτικές της. Προς τα έξω πουλάει την ειρήνη. Αλλά αυτό αποτελεί απλώς μια φορμή για να ε, χρηματοδοτηθούν ε, μόνο στρατιωτικέ αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων τρίτων χωρών. Η δεξιά και η σοσιαλδημοκρατία προσπαθούν να επιβάλλουν ένα πολεμοχαρές πνεύμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που προωθεί την, τον πόλεμο και δεν υπερασπίζεται την ειρήνη. Η υπεράσπιση της ειρήνης περνάει από την διάλυση του ΝΑΤΟ ή των στρατιωτικών δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ε, λέει και η βάση την οποία στηρίχθηκε η σύγχρονη δημοκρατία της Πορτογαλίας. Θα πρέπει να γίνεται σεβαστή η χάρτα των Ηνωμένων Εθνών και τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πιμέντα Λόπες. Κάτσε διάει τρεις συνάδελφοι. Η κυρία Ward πρώτη. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καταρχήν ένα όραμα ειρήνης. Να σας υπενθυμίσω επίσης ε, την έκκληση ειρήνης των Βρυξελών που, που ήταν αποτέλεσμα μιας, ενός συνεδρίου για την ευημερία και την ειρήνη στις 28 Νοεμβρίου του 2011 εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή η δήλωση προθέσεων είχε ως στόχο να ενθαρρύνει σχέδια και δράσεις που θα προωθούν την ειρήνη στο, με, τον, με την παγκόσμια έννοια τη, που θα εμπνέεται από την ανθρώπινη εξηρότητα, την ελευθερία, την ισότητα και την αλληλεγγύη, όπως αναφέρονται στο προήμιο των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν επιβεβαιωθεί και από τη Συνδική της Λισαβόνας το 2009. Το βραβείο Νομπέλ για την ειρήνη που δόθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραμμίζει τη σημασία αυτών των δράσεων, μεταξύ αυτών και τη δήλωση προθέσεων. Η δήλωση αυτή προθέσεων είχε ως στόχο να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για να ξεκινήσει μια σειρά δράσεων για να οικοδομηθεί ένας κόσμος ευμερίας και ειρήνης και θα πρότεινα η επόμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υπογράψει ε, την εκκλησία αυτή και να προβεί σε δράση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φλάναγκα